μας ε, ε, δεν θα το καθορίσουν αυτοί που είναι πιο βραδείς ε, και βρίσκονται σε υστέρηση, αλλά πιο γενναιόδοροι και οι πιο φιλοευρωπαϊστές. Αυτοί θα καθορίσουν την ατζέντα μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ συνάδελφε Θέρκας. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Θα γίνει η, η ψήφιση αύριο στις 12 το μεσημέρι. Επόμενο θέμα είναι προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την εγγύηση για την νεολαία για την απασχόληση και κοινωνικά ε, ζητήματα. Καταρχήν, ως συντάκτρια της ερώτησης, η κυρία Πεβάνς Μπερές θα λάβει τον λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, από τον Ιούλιο υποβάλλεται μία πρωτοβουλία για μία εγγύηση για τους νέους πρωτοβουλία που σας είχε ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και έκτοτε τα πράγματα έχουν εξελιχθεί και στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργών Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης στις 7 και 8 Φεβρουαρίου του 2013 στο Δουβλίνο θα πρέπει να συζητήσει την πρωτοβουλία αυτή. Έχουμε υποβάλει αυτή την προφορική ερώτηση και θα εγκρίνουμε και ένα ψήφισμα προκειμένου να στηρίξουμε κάθε σχετική πρωτοβουλία και κάθε σχετικό μέτρο το οποίο θα υποστηρίξει αυτή την εγγύηση για τους νέους. Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία για τους νέους στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προωθηθεί. Η υφιστάμενη κατάσταση απασχόληση των νέων είναι απαράδεκτη. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στην Αυστρία, τη Σουηδία, στη Δανία, αλλά ακόμα και στην εγγύηση αυτή που υφίσταται στη Γαλλία. Υπάρχουν ουσιαστικά κάποιες χώρες οι οποίες έχουν εγκρίνει σχετικές νομοθεσίες και θα πρέπει να θεωρούμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μπορεί να υπάρξει μια ξεχωριστή νομοθεσία υποστήριξης των νέων. Δεν μπορεί ένας νέος να βρίσκεται χωρίς δουλειά ή να βρεθεί, να βγει από το σύστημα μόρφωσης, κατάρτισης, χωρίς να μπορεί μέσα σε τέσσερις, σε τέσσερις μήνες να βρει κάποιο άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, εκπαίδευσης ή μία εργασία. Δεν θέλουμε να υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν θέσει εργασία. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι να δημιουργηθούν όλε τι απαραίτητε ευκαιρίε προκειμένου να μην χαθεί αυτή η γενιά. Κάνατε λοιπόν μια πρόταση η οποία βασίζεται πάρα πολύ στην καλή βούληση και θέληση των κρατών μελών. Ουσιαστικά τους δίνεται δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα διαφορετικά ταμεία και ιδίω το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ζήτημα επί του οποίου χρειάζεται και η δική μας σύμφωνη γνώμη. Εμείς θέλουμε η πρόταση αυτή να είναι ρεαλιστική. Πρέπει όμως να πούμε και προς τα κράτη-μέλη ότι αν πραγματικά θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε αυτή την πρωτοβουλία, την εγγύηση για τον νέο, χρησιμοποιώντα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τότε θα πρέπει να είμαστε συνεκτικοί και συνεπεί και θα πρέπει να επιτρέψουμε ένα 25% του υφιστάμενου ποσού τη πολιτική συνοχή να δοθεί υπέρ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Πρέπει επίσης, κατά την άποψή μου, να εξετάσουμε τα πράγματα πέρα από την πρωτοβουλία αυτή και να δούμε πώς θα καταφέρουμε να εξορροπήσουμε τις μακροοικονομικές ανισορροπίες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να καταφέρουμε να κάνουμε την πρωτοβουλία αυτή εγγύηση των νέων μια πραγματική ευρωπαϊκή πρόκληση που θα υποστηρίζεται από πραγματικά ευρωπαϊκά μέσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ασχοληθεί το Συμβούλιο του Φεβρουαρίου με το ζήτημα αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Επίτροπε, επιθυμεί η εγγύηση αυτή για τους νέους να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα την οποία βιώνουν οι νέοι σε κάθε χώρα. Γιατί δεν πρόκειται μόνο βέβαια για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλάμε. Πολύ συχνά τα πιο ευάλωτε ομάδε στα πλαίσια του πληθυσμού αυτού του άνεργου είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την ευρωπαϊκή υπηκότητα. Άνθρωποι που είναι θύματα στιγματισμού ακόμα περισσότερο επειδή είναι άνεργοι. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε του ανθρώπου αυτού γιατί διαφορετικά προτιμάζουμε ένα πρόσφορο έδαφο για όλου αυτούς, ε, για όλες αυτές τις λαϊκιστικές ε, τάσεις που βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε επίση αυτή η εγγύηση για τους νέους να λάβει υπόψη της ε, την πραγματικότητα, την πραγματική κατάσταση στην οποία αντιμετωπίζουν οι πτυχιούχοι. Γιατί ξέρετε ότι για τους περισσότερους η πρόσβαση στην αγορά εργασίας είναι πάρα πολύ δύσκολη και βέβαια δεν επιτυγχάνεται στα 25 έτη. Την προηγούμενη εβδομάδα, σε σχέση με μια έκθεση για την απασχόληση των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπατε κι εσεί ότι ένα πέπτο των νέων σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν δουλέψει ποτέ και τα τρία τέταρτα βρίσκονται κάτω των 35 ετών. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να λάβουμε υπόψη μα τα δεδομένα αυτά, αν δεν θέλουμε όχι μόνο αυτή η γενιά να χαθεί, αλλά αν θέλουμε όντω η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη, να καταφέρει να ανταποκριθεί στην σημαντική αυτή πρόκληση, στην πρόκληση της καινοτομία. Γιατί ποιος μπορεί να εγγυηθεί την καινοτομία καλύτερα από νέους οι οποίοι εκπαιδεύονται, καταρτίζονται και εργάζονται. Μόνο η νεολαία τελικά μπορεί να μα επιτρέψει να βρεθούμε στην αιχμή του δόρατο όσον αφορά την τεχνολογική πρόοδο και την κοινοτομία. Μόνο οι νέοι μπορούν να εγγυηθούν το μέλλον και τι αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο οι νέοι μπορούν να προωθήσουν και να εγγυηθούν το μέλλον του κοινωνικού μοντέλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είχε πει και ο πρόεδρο Μπαρόσο πριν από λίγο καιρό. Κύριε Επίτροπε, ξέρετε ότι εμεί κατά τη διάρκεια του επόμενου Συμβουλίου Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόληση θα ασκήσουμε την κατάλληλη πίεση προκειμένου η πρόταση αυτή να γίνει πραγματικότητα. Σα ευχαριστούμε πολύ αγάπητη συνάδελφε κυρία Μπερέ. Ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Επίτροπε Άντορα, έχετε τον λόγο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, με βουλευτές θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων που κατέθεσε το προφορικό αυτό ερώτημα και την πρόταση ψηφίσματο, γιατί δείχνει την ε, μεγάλη αφοσίωση του Κοινοβουλίου στην πρόταση αυτή για τη δημιουργία μια εγγύηση για την όλη. Θα ήθελα να μιλήσω ε, πιο αναλυτικά για κάποια θέματα. Πρώτα απ' όλα συμφωνώ με την κυρία Μπερέ ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Είναι κρίσιμη η εγγύηση για την όλα σίγουρα έχει ένα οικονομικό κόστος, αλλά το κόστος της αδράνειας θα είναι πολύ ψηλότερο και η ανεργία η νεανική είναι πάρα πολύ δαπανηρή γιατί κοστίζει 150 δις ε, ετησίως στην Ευρώπη ενώ υπάρχει απώλεια σε εισοδήματα και σε ε, φορολογικά έσοδα σύμφωνα με το Ίδρυμα Eurofound. Επίσης ε, υπάρχει ένα μεγάλο κόστος και της μακροχρόνιας ανεργίας όχι μόνο για την οικονομία αλλά και για την κοινωνία, ανησυχία για την νεολαία, μέλλον δύσκολο, κοινωνικός αποκλεισμός ενδεχομένως, φτώχεια. Η εγγύηση για την όλη λοιπόν είναι μια επένδυση. Γι' αυτό και η Επιτροπή θα διαθέσει περαιτέρω κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αλλά και από τα άλλα διαρθρωτικά ταμεία. Τα ακριβή ποσά, όπως ξέρετε, θα εξαρτηθούν από την έκβαση των διαπραγματεύσεων για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Επομένως, βασιζόμαστε στη δική σας υποστήριξη για να έχουμε ένα ισχυρότερο κοινωνικό ταμείο την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Επίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλι ξεκίνησε διαπραγματεύσει με τα κράτη-μέλη για το περιεχόμενο των συμφωνιών εταιρική σχέση και των επιχειρησιακών προγραμμάτων για την περίοδο 2014-2020. Θέλουμε λοιπόν να επικεντρωθούμε στη μετάβαση από το σχολείο στην εκπαίδευση. Έχουμε διαπραγματεύσει λοιπόν και θα συζητήσουμε και τα ποσά που θα διατεθούν για τέτοιου είδου σκοπού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί απόλυτα ότι προκειμένου αυτά τα σχήματα να είναι αποτελεσματικά θα πρέπει να υπάρχουν ε, ισχυρές εταιρικέ σχέσεις μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων. Αντιλαμβανόμαστε όμως ταυτόχρονα ότι δεν είναι εύκολο αυτό για ορισμένα κράτη-μέλη και θα πρέπει να βασιστούμε στην εμπειρία που έχουν αναπτύξει κράτη-μέλη που ήδη έχουν τέτοια σχήματα. Προτείνουμε λοιπόν έξι συγκεκριμένε συστάσει που θα αποτελέσουν κατευθυντήριε γραμμέ για την συμπήξη τέτοιων ισχυρών εταιρικών σχέσεων. Επίση, η ε, προσπάθεια που ξεκίνησε το καλοκαίρι ε, με προπαρασκευαστική δράση επικεντρώνεται στην θέσπιση και συγκρότηση αυτών των ε, εταιρικών σχέσεων και περιμένουμε πώς θα ολοκληρωθεί ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα επιλεγεί το project τι επόμενε εβδομάδε και βέβαια θα υπάρξει ανταλλαγή των γνώσεων και των καλών πρακτικών με όλα τα κράτη-μέλη. Έχουμε επίγνωση ω Κομισιόν των περιορισμών ότι υπάρχουν μέτρα λιτότητα, ιδίω ε, σε κράτη που έχουν οξέα προβλήματα, μεγάλη ανεργία, ιδίω μεταξύ των νέων. Θα επαναλάβω όμω ότι θα έχουμε θετική επιστροφή από την επένδυσή μα σε αυτή την εγγύηση για την νεολαία. αναφέρουμε και το δείχνει και η ετήσια έρευνα για την ανάπτυξη έθεση το 2013, αλλά και η ανακοίνωση Κομισιόν για την ποιότητα των δημοσίων δαπανών. Εκεί η εγγύηση για την νεολαία ε, θεωρούνται μέτρα πάρα πολύ θετικά. Σίγουρα βέβαια η προσέγγιση δεν θα πρέπει να είναι ε, η ίδια για όλες τις περιπτώσεις. Ε, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την πολυμορφία, τα διαφορετικά σημεία κίνηση σε ό,τι αφορά την ανεργία των νέων, ή τη δυνατότητα των φορέων ε, τη αγορά εργασία σε κάθε κράτο μέλο. Επίση, οι νέοι που είναι ο στόχο αυτών των ε, σχημάτων, αυτών των μηχανισμών, δεν είναι ομοιογενή ομάδα. Και εκτό αυτών, θα πρέπει κάθε κράτο μέλο να δει και τις ε, διαφορετικές ανάγκες ορισμένων ομάδων. Υπάρχουν ομάδε νέων που αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια για την είσοδο στην αγορά εργασία. Πάντω. Πρέπει να υπάρξει μια έντονη ευρωπαϊκή διάσταση γιατί είναι κοινό ο στόχο τη στήριξη τη νεολαία. Πρέπει λοιπόν να καταδείξουμε την αλληλεγγύη μα, ιδίω ε, σε αυτού του ε, καιρού τη μεγάλη νοσονομική λιτότητα, χωρί όμω ε, να διακυβεύσουμε το μέλλον μα όταν προσπαθούμε να παγιώσουμε κάπω την οικονομική κατάσταση και να εξηγιάνουμε τα οικονομικά. Θέλουμε να υπάρξει πολυμερή εποπτεία επίση ε, για την ε, εγγύηση για την νεολαία, τα σχετικά σχήματα και έχουμε και το πρόγραμμα τη αμοιβαία μάθηση ε, Mutual Learning, ώστε να υπάρξει μια ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των κράτων μελών. Θα το ενθαρρύνουμε αυτό. Επίση θα παρακολουθούμε τακτικά και θα αναφέρουμε σε σχέση με τι εξελίξει για την μελέτη, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη χρήση αυτών των εγγύσεων για την νεολαία στο πλαίσιο του ετήσιου ε, προγράμματος για τις δημόσιες ε, νομικές υπηρεσίες και θα έχουμε και σημαντική ε, συνεισφορά στη δημιουργία αυτών των εταιρικών σχέσεων. Τέλος, θέλω να σας ενημερώσω ότι ήδη είχαμε μια πρώτη παρουσίαση της πρότασης για την εγγύηση για την νεολαία στις 18 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Πολλά κράτη-μέλη χαιρέτησαν θερμά αυτή την πρωτοβουλία και υποσχέθηκαν να εργαστούν επικοδομητικά προς την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας της 28 ε, Φεβρουαρίου, οπότε και θα συνεδριάσω στο Συμβούλιο ε, Κοινωνικών Υποθέσεων Πλανητικής Πρεδέσης, παραλαμβάνω. Σας ευχαριστούμε, Επίτροπε Άντορ. Οι αγορητές εξωμένως των ομάδων. Ο κύριος Έρη, δύο λεπτά, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ΕΛΚ, και η ομάδα Ευρωβουλευτών του ΕΛΚ αυτή την πρωτοβουλία την έχει ήδη χαιρετήσει και καλωσορίσει. Θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση είναι θετική, πολύ θετική και γνωρίζουμε τα σχετικά γεγονότα και στοιχεία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ανεργία των νέων είναι σχεδόν, αυξήθηκε κατά 23 σχεδόν σε 100 Έχουμε εκατομμύρια νέου σήμερα που δεν έχουν δουλειά στις χώρες μας. Σε κάποιες χώρες είναι 25% το ποσοστό ανεργία των νέων και σε κάποιες χώρες μάλιστα και 45% το ποσοστό ανεργία των νέων. Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα, να αλλάξει αυτή η κατάσταση πραγμάτων. Και γι' αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργά δραστηριοποιείται σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Όμως θα πρέπει από την άλλη πλευρά και να αναγνωρίσουμε όταν θέτουμε το ερώτημα ποιος θα πληρώσει το κόστος στις δαπάνες αυτών των προγραμμάτων. Παραμένει το ερώτημα, δεν έχουμε σαφή απάντηση αυτού του ερωτήματος. Βρισκόμαστε σε ένα πεδίο αβεβαιότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες. Βλέπουμε όμως ότι επανειλημμένα, ας το πω εσύ χρησιμοποιούνται αυτά τα κονδύλια προς αυτή την κατεύθυνση σε πολλές περιπτώσεις αφήνονται, εγκαταλείπονται τα κράτη-μέλη και μένουν μόνα τους. Πρέπει να αλλάξει η κατάσταση πραγμάτων. Η κατάσταση σε σχέση με τα διάφορα κράτη-μέλη, σε σχέση με την ε, διαμόρφωση των ποσοστών ανεργίας, βλέπουμε ότι είναι διαφορετική κατάσταση από χώρα σε χώρα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε διαφοροποιημένες προτάσεις που θα λαμβάνουν υπόψη αυτές τις ιδιομορφίες. Θέλω να τονίσω ότι δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνη της ε, που μπορεί να δημιουργήσει αυτές τις θέσεις απασχόλησης, αλλά μια δυναμική εν συνόλο οικονομία στο σύνολό της. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής που πρέπει να διευρυνθούν για να είναι πιο αποτελεσματικά. Ευχαριστούμε κύριε Έρη. Ο κύριος Θέρκας, τώρα ένα λεπτό παρακαλώ. Μικρόφωνο. Μικρόφωνο παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, οι σοσιαλιστές βουλευτές είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την πρωτοβουλία. Έχετε τη στήριξή μας στην απόλυτη και ελπίζουμε στο Συμβούλιο Εύσκο να δοθεί συνέχεια στην εξαιρετική αυτή ιδέα. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Ακούμε πολλέ φορέ να γίνεται λόγο για το 50% των ε, νέων ανέργων. Αλλά υπάρχουν μέση όροι ε, και υπάρχουν και συγκεκριμένε περιοχέ, όπω η δική μου περιοχή, που φτάνει η ανεργία το 65% ή το 70% ή σε άλλε περιοχέ φτάνει το 80% η ανεργία των νέων. Είναι ε, πραγματικότητα. Δεν μιλάμε τελικά απλά για ένα πρόβλημα, για μια τραγωδία. Και πραγματικά, όπω το μέλλον των νέων, το δικό μα μέλλον, πρέπει να το εγγυηθούμε. Και θα πρέπει να γίνει μια αλλαγή ε, στα κράτη-μέλη, γιατί τα κράτη-μέλη ε, έφεραν την τραγωδία με αυτά που έκαναν μέχρι τώρα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν φάνταστα μέτρα, ε, να ε, συνεργαστούν όλοι οι κοινωνικοί εταίροι, γιατί δεν είναι πρόβλημα μόνο των νέων, αλλά όλων μας αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε Θέρκας. Για δύο λεπτά η συνάδελφος κυρία Χίρς παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, για την ανεργία των νέων που είναι πάνω από 20% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κάποιες χώρες και πάνω από 50% δεν είναι θέμα πλέον ότι πρέπει αμέσως να δραστηριοποιηθούμε. Δεν το συζητούμε αυτό και όχι με μέτρα που μετά από χρόνια θα έχουν αποτελέσματα, αλλά με μέτρα που άμεσα θα προσφέρουν δυνατότητες να έχουν νέες προοπτικές αυτοί οι άνεργοι νέοι. Γι' αυτό υποστηρίζουμε εμείς οι φιλελεύθεροι την ε, προσπάθεια, την πρωτοβουλία της εγγύησης των, για τους νέους. Δεν θέλουμε να χαθεί μια γενεά νέων. Επιπλέον όμως ε, μια τέτοια εγγύηση για την νεολαία δεν μπορεί να είναι εγγύηση για την απασχόληση. Οι θέσεις απασχόλησης δημιουργούνται από την οικονομία. Δεν μπορούμε εμείς να τις δημιουργήσουμε με μέσω ενός προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα μαγικό ραβδί. Όμως, μια ευρωπαϊκή εγγύηση μπορεί να βοηθήσει τους νέους. Αυτά που υπάρχουν σήμερα να διευκολυνθούν, να διευκολυνθεί η πρόσβαση των νέων, τα προσκόμματα να αντιμετωπιστούν. Στην αρχή του έτους ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα στην Γερμανία για παράδειγμα. Το πρόγραμμα στην, για την υποστήριξη και προώθηση της κινητικότητας των νέων ώστε να μπορέσουν στην Ευρώπη άτομα με προσόντα να μπορέσουν να ε, προωθηθούν και να υποστηριχθούν και εκείνοι που δεν έχουν θέση απασχόλησης να μπορέσουν να προσθέσουν στη Γερμανία και να βοηθηθούν. Εδώ οι πρωτοβουλίε από τα κράτη-μέλη πρέπει να συνδυαστούν με μια εγγύηση για την νεολαία, ευρωπαϊκή εγγύηση. Αυτή η ευρωπαϊκή εγγύηση μπορεί μόνο μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου να χρηματοδοτηθεί. Εκεί υπάρχουν τα κονδύλια. Τώρα μπορεί η Ευρώπη να δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι υπάρχει δυναμικό για την ευρωπαϊκή αγορά εργασία για του νέου και μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση, αυτόν τον προσανατολισμό, ώστε στο μέλλον να έχουν προοπτικέ αυτοί οι νέοι. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πολύ πολύ συνάδελφε Χίες. Ακολουθεί η συνάδελφος κυρία Τούρουνεν. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Η κατάσταση των νέων στην Ευρώπη υπό κάθε πρίσμα είναι πολύ αρνητική. Είναι πάρα πολλοί οι νέοι που δεν έχουν εργασία και οι οικονομικές τους προοπτικές είναι αρνητικές. Εμείς ως Ευρωπαίοι πολιτικοί, υπεύθυνοι Ευρωπαίοι πολιτικοί, πρέπει να διαρωτηθούμε και να δούμε μήπως χάσουμε μια ολόκληρη γενεά και τη θυσιάσουμε. Πρέπει να μεριμνήσουμε η νέα γενεά να υποστηριχθεί και να διαφυλαχθεί και από την αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να μην έχει αυτή η νέα γενεά χειρότερες ή αρνητικότερες προοπτικές από ότι οι γονείς μας. Οι γονείς μας, η μητέρα μου όταν ήταν νέα στη δεκαετία των 80 έδωσε αγώνα για την, ε, να μπορέσει να ε, βρει εργασία στην αγορά εργασίας. Από τη δεκαετία του 80 γνωρίζουμε ότι η ανεργία των νέων έχει πάμπολα αρνητικά χαρακτηριστικά και συνεπάγεται πολλά αρνητικά στοιχεία για τους νέους. Πρέπει μάθουμε από τα σφάλματα του παρελθόντος επιτέλους και πρέπει με σθένος να δράσουμε ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε μέσω της εγγύησης για την νεολαία, ευρωπαϊκή εγγύησης. Το παράλογο εδώ είναι ότι οι νέοι στην Ευρώπη βρίσκονται σε μια απελπιστική που δημιουργεί απόγνωση ανεργία και που έχουμε ε, πραγματικά ευθύνες που πρέπει να υπομισθούμε. Ε, είναι μια παράδεκτη κατάσταση η ανεργία των νέων. Η εγγύηση για την νεολαία είναι μια θετική πρωτοβουλία σε μια οικονομική περίοδο κρίσης. Υπέβαλε πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευχαριστούμε γι' αυτό. Τώρα είναι η μπάλα στο Συμβούλιο και στην Ιρλανδική Προεδρία. Εκείνη πρέπει να πράξει κάτι. Έχουμε υψηλότατες προσδοκίες όπως και οι Ευρωπαίοι πολίτες συνολικά. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε συνάδελφε κυρία Τουρούνεν. Ακολουθεί για 1,5 λεπτό ο συνάδελφο Λε Ιαρίκ, παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, κύριε και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να αποτελεί πλέον όρο συνώνυμο με την ανεργία. Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα χιλιάδες νέου που καλύπτει η εγγύηση των νέων θα πρέπει ουσιαστικά να υποστηριχθεί. Θα πρέπει να υποστηριχθεί η πρωτοβουλία αυτή όχι ω κοινωνικό μέτρο αντιμετώπιση ανεργία, αλλά ω ένα κοινωνικό μέσο συνεργασία, για να προσφέρουμε ένα μέλλον στους νέους. Για να θυσιάσουμε τις νέες γενιές των νέων είναι τελικά η καλύτερη εγγύηση για την κατάρρευση, την αυριανή κατάρρευση της Ευρώπης. Θεωρώ ότι υπάρχει κάτι παράλογο στην πολιτική που ακολουθούν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιέζουν πάρα πολύ για την αύξηση του ορίστου ταξιοδότησης, ενώ αφήνουν πάρα πολλούς νέους χωρίς εργασία. Η πρωτοβουλία εγγύηση για του νέου θα πρέπει να συνοδεύεται από νέα δικαιώματα. Δικαίωμα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη μόνιμη εκπαίδευση και κατάρτιση. Θα πρέπει επίση να δίνονται δεύτερε ευκαιρίε, νέε ευκαιρίε, όπω επίση και το δικαίωμα να συνδικαλιστούν οι νέοι αυτοί. Τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει να είναι καθολικά, να ισχύουν για όλους τους Ευρωπαίους και να επίση εξασφαλίζουμε στου νέους αυτούς ένα ισότιμο ελάχιστο μισθό, μια απαραίτητη κοινωνική υγειονομική κάλυψη, πρόσβαση επίσης στα συστήματα περίθαλψης και θα πρέπει να προβλέπονται τα παράλληλα κατάλληλα προγράμματα τα οποία θα συνδυάζουν την εργασία με τα προγράμματα κατάρτιση. Η θέσπιση λοιπόν της εγγύησης για τους νέους θα πρέπει να λάβει χώρα με ένα ταμείο το οποίο θα χρηματοδοτεί την πρωτοβουλία αυτή, ξεχωριστό ταμείο και όχι με μετάθεση. Ε, Σας ευχαριστούμε συνάδελφε η Λέη Αρίκα. Αυτοί ήταν οι αγορητές των ομάδων. Τώρα έχουμε τους άλλου ατομικά εγγεγραμμένους. Μαν, 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα και την Ισπανία είναι απαράδεκτα υψηλή. 45% στην πατρίδα μου τη Γερμανία χαμηλότερο ποσοστό. Μια δραματική κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε οδηγασμό, κατακαιρματισμό της Ευρώπης και σε μια θυσιασμένη, χαμένη γενεά. Είχαμε ένα πακέτο πρόσφατα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που το καλοχαιρετίζουμε ο πυρήνα τη εγγύηση για τους νέους ήταν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν προτείναμε σε μια έκθεση να υπάρξει η ε, δικαιοσύνη έναντι των γενεών. Μια ε, δίκαια συμφωνία, ένα σύμφωνο δικαιοσύνης μεταξύ των γενεών. Δεν, ε, ήταν, δεν κατάφεραν να, να αποκτήσουν κάποιοι προσόντα και επαρκή προσόντα για την, ε, το επάγγελμά τους. Ε, θα πρέπει να βοηθηθούν. Αυτή η εγγύηση με βάση το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο βασίζεται στην ε, βάση στα θεμέλια της προώθησης και έτσι θα προτείνονται μέτρα τα οποία θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά ώστε να βοηθηθούν οι νέοι. Ας αποφύγουμε την περιθωριοποίηση των νέων. Καταρτισμένοι με δεξιότητες νέοι μπορούν να συνεισφέρουν ε, για την ευδοκίμηση των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Πρέπει να επενδύσουν τα κράτη περισσότερα για την κατάρτιση. Έχουμε χώρες ε, όπως τη Γερμανία που έχουμε το διτό σύστημα εκπαίδευσης. Ε, υποστηρίζουμε με μια χρηματοδότηση έναξης με 10 εκατομμύρια ευρώ αυτό το ελπιδοφόρο κίνημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ακολουθεί Ρέγνερ παρακαλώ στη συνέχεια. Η κυρία Ρέγνερ, σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, γνωρίζετε τα αριθμητικά στοιχεία πολύ καλά. 5,5 εκατομμύρια νέοι είναι άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. 56,6% είναι το ποσοστό ανεργίας των νέων στην Ισπανία. Δεν είναι μόνο αριθμητικά στοιχεία, είναι ένα σκάνδαλο αυτό πρέπει πραγματικά να δράσουμε με πολλά θαυμαστικά μετά από αυτή την ε, ε, διακήρυξη. Έχουμε το πρόγραμμα καταπολέμησης ανεργίας των νέων. Χαιρετίζουμε το πακέτο μέτρων που προτάθηκε και παρουσιάστηκε στις 5 Δεκεμβρίου. Προέρχομαι από την Αυστρία, μια χώρα που με την εγγύηση για την κατάρτιση δίνει ένα από τα καλύτερα παραδείγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Έχουμε το διτό σύστημα κατάρτισης. Ε, εκτιμούμε ιδιαίτερα την κοινωνική εταιρική σχέση για την αντιμετώπιση της ανεργία. Είναι μια ε, συνταγή επιτυχίας. Όμως ε, δεν πρέπει να το ε, παρασιοποιήσουμε. Πολλά χρήματα απαιτούνται. Και αν το κάνει τώρα η Ελλάδα ή η Ισπανία θα πρέπει ευρωπαϊκά να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί όχι για παράδειγμα να υπάρξει ένα ξεχωριστό ταμείο για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Γιατί να μην έχουμε τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που θα πρέπει να μετατεθούν και να χρησιμοποιηθούν και για νέους στόχους. Θέλω ένα παράθεμα να ολοκληρώσουμε ολοκληρώσω. Διακόπτει ο πρόεδρο. Συνάδελφε, λυπούμε πολύ. Έχετε ξεπεράσει τον χρόνο. Πρέπει κάπω να είμαστε πιο πειθαρχημένοι. Παρ' όλα αυτά σα ευχαριστώ. Στη συνέχεια η συνάδελφο Χάρκιν. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω την πρόταση για την εγγύη για την Ολέα και αν εφαρμοστεί θα είναι ένα απτό ε, δείγμα του ότι αντιδράει η Ευρώπη. Είναι όμως ένα μικρό βήμα και είναι ένα πρώτο βήμα. Και πρέπει να δούμε και την ευρύτερη εικόνα ότι πολλές χώρες ε, μειώνουν ε, τις κοινωνικές, μάλλον, τις κοινωνικές επενδύσεις λόγω των αυστηρών προγραμμάτων λιτότητας που συνεχίζουν να εφαρμόζουν. Και στην Ιρλανδία έχουμε 29,7% ανεργία των νέων. Δεν είναι η χειρότερη βέβαια, αλλά τα πραγματικά ποσοστά νομίζω είναι υψηλότερα. 87.000 νέοι κυρίως Ιρλανδοί εγκατέλειψαν τη χώρα γιατί δεν έβρισκαν δουλειά στη χώρα. Ο πρόεδρος Χίγκιν στην προηγούμενη χρονιά είπε ότι έχω επίγνωση ε, της ε, διαφωνίας αυτής του, και της της αντίφασης που υπάρχει ε, που ε, έχω ασχοληθεί με όλα αυτά. Υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό που είναι άνεργοι και ξέρουμε ότι σε κάποιες χώρες 55% των νέων είναι άνεργοι και πρέπει να μην την παραγνωρίζουμε αυτή την πραγματικότητα. Το είπατε και εσείς, δεν θα πρέπει να δεσμεύσουμε το μέλλον μας όταν προσπαθούμε να εξηγιάνουμε τα οικονομικά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε Χάρκιν. Ακολουθεί η κυρία συνάδελφος Σρόιτερ. Ένα λεπτό παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το Συμβούλιο με μεγάλες διακηρύξεις θεωρεί ότι η ανεργία των νέων είναι το μέγιστο πρόβλημα της κρίσης. Τώρα αναμένουμε μετά από αυτά τα λόγια να ακολουθήσουν πράξεις αξιόπιστη θα είναι μόνο μια δεσμευτική εγγύηση για τους νέους. Δηλαδή ένα δικαίωμα το οποίο θα μπορούν να διεκδικήσουν οι νέοι σε κάθε κράτος μέλος. Και φυσικά συγκεκριμένα μέτρα, δηλαδή προσφορά κατάρτισης και εργασίας για τους νέους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει με μηχανισμούς αξιολόγησης κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αυτή την εγγύηση για τους νέους να την διασφαλίσει, να την κατοχυρώσει στα κράτη-μέλη. Απευθύνουμε έκκληση και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναμένουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από τα λόγια να ακολουθήσουν πράξεις εμείς ε, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποβάλαμε προτάσεις ε, για υποστήριξη, για καινοτομία και μέσω των κονδυλίων ε, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που θα βοηθήσουν τους νέους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Με αυτές τις προτάσεις όμως αντιμετωπίζουμε αντιστάσεις. Αντιστάσεις και σε σχέση με την, με την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ζητούμε από την Επιτροπή και εκπροσώπηση της Επιτροπής μετά από τα λόγια που ε, μας εξέθεσαν να ακολουθήσουν οι πράξεις και να είναι συνεπεί στι πράξει του. Σα ευχαριστούμε κυρία Σρόιτερ. Για 1,5 λεπτό ο κύριο Πουπάκη παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Οι νέοι σήμερα αποτελούν τα μεγαλύτερα θύματα τη κρίση, γι' αυτό και η νεανική ανεργία σαν κορυφαίο πρόβλημα απαιτεί πλέον άμεσε και δυναμικέ παρεμβάσει. Στη χώρα μου την Ελλάδα το 56% των νέων είναι εκτό αγορά εργασία, με ιδιαίτερα επώδυνε επιπτώσει τόσο στη δική του ζωή όσο και συνολικότερα στη λειτουργία τη κοινωνία. Κύριε Επίτροπε, θεωρώ ότι είναι χρέο όλων μα να εγγυηθούμε ότι οι νέοι Ευρωπαίοι δεν θα γίνουν μια χαμένη γενιά. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μοχλό πίεση προ τι κυβερνήσει, του κοινωνικού εταίρου και του άλλου εμπλεκόμενου φορεί, ώστε να υιοθετήσουν στοχευμένε δράσει, χωρί όμω να λειτουργήσουν σε βάρο άλλων πολιτικών κοινωνικού χαρακτήρα. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, σε μια περίοδο εκτεταμένων περικοπών στου εθνικού κοινωνικού προπολογισμού και στα εκπαιδευτικά κονδύλια, με πιο συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένα μέτρα μπορείτε να διασφαλίσετε ότι η εγγύηση για τους νέους θα χρηματοδοθεί αλλά και θα εφαρμοστεί αποτελεσματικά στα κράτη μέλη ιδίως σε αυτά μάλιστα που υπάγονται σε καθεστώς μνημονίων. ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ συνάδελφε Πουπάκη. Για ένα λεπτό η κυρία Κοστέλο παρακαλώ τώρα. Κύριε Πρόεδρε, Είμαι υπέρ των προτεραιοτήτων της Ιρλανδικής Προεδρίας όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση. Παρ' όλα αυτά, οι προκλήσεις είναι πολύ σημαντικότερες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι η πρόταση αυτή θα πρέπει να αποτελέσει το πιο σημαντικό σημείο της συζήτησης του Συμβουλίου που θα γίνει το Φεβρουάριο στην Ιρλανδία. Έχουμε ποσοστά της τάξης 33% στην Ιρλανδία και βρισκόμαστε στην, στο πέμπτο μεγαλύτερο ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά έχουμε χάσει μια γενιά. Πάρα πολλοί άνθρωποι μένουν άνεργοι ή καταφεύγουν στο εξωτερικό. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Ιρλανδία ο πρόεδρος Μπαρόσο αναφέρθηκε στην εγγύηση των νέων στα πλαίσια του διαλόγου που έλαβε χώρα εκεί. Η ιδέα αυτή, η πρωτοβουλία αυτή έγινε δεκτή από τους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση αυτή. Ωστόσο, αν πραγματικά θέλουμε την εγγύηση για τους νέους, χρειαζόμαστε και την απαραίτητη χρηματοδότηση όπως είπε η κυρία Μπερέσα. Πρέπει να καταφέρουμε να στείλουμε ένα μήνυμα για δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα αυτό. Τέλος, κύριε Επίτροπε, όσον αφορά τα, πολιτι... τα πιλωτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς αυτά θα λειτουργήσουν στην Ιρλανδία, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα το οποίο προβλέπετε. Σας ευχαριστούμε πολύ συνάδελφε κυρία Κοστέλο. Για ένα λεπτό η κυρία Ντέλη παρακαλώ. Είναι επίγον κύριε Επίτροπε. Μια ολόκληρη γενιά θυσιάζεται στο βωμό της λιτότητας. 14 εκατομμύρια νέων κάτω από τα 30 ούτε θέση εργασίας έχουν ούτε είναι στις σπουδέ, αλλά λέμε ότι υπάρχει λύση. Εδώ και χρόνια οι πράσινοι προτείνουν την εγγύηση για την ολέα στην Αυστρία, στην Δανία και σε άλλες χώρες Δύο είναι οι προθέσει που χρειάζονται για να λειτουργήσει. Πρώτον, θα πρέπει να έχουμε ένα πραγματικό εισόδημα αυτονομία, αυτάρκεια, γιατί πολλοί νέοι εργάζονται όσο σπουδάζουν και πολλέ φορέ αποτυγχάνουν σπουδέ του λόγω αυτού. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχουν σαφεί κανόνε που θα πλαισιώνουν τι περιόδου άσκηση. Η Κομισιόν δεν μπορεί να περιμένει άλλο για να καταπολεμήσει πλέον την εκμετάλλευση των νέων οι οποίοι ε, προσλαμβάνονται σε ε, κάποια θέση που δεν είναι όμω σε καμία περίπτωση ασκούμενοι, αλλά έχουν ένα ε, ορισμένου χρόνου συμβόλαιο και πρέπει να γίνει μια ε, επένδυση στην νεολαία για να δώσουμε ελπίδα στους νέους. Είναι όμως μια πρόκληση για όλους μας σήμερα, γιατί πρέπει να επανασυμφιλιώσουμε τους νέους με την Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Αντέλη για μισή λεπτό η κυρία συνάδελφος, η κυρία Μπάστος παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινάμε τη χρονιά με επίπεδα ανεργίας δραματικά υψηλά. Στην χώρα μου την Πορτογαλία έχουμε φτάσει στο υψηλότερο ποσοστό της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη και ζούμε ένα κύμα μετανάστευσης ε, παρόμοιων διαστάσεων όπως είχαμε κατά τη δεκαετία του 60 τον προηγούμενο αιώνα. Αυτό το κύμα θα έχει επιπτώσεις και έχει επιπτώσεις κυρίως στους εκπαιδευμένους νέους ε, για την αναζήτηση εργασίας αναζητούν επαγγελματικά μια διέξοδο εκτός της χώρας μας αυτή η νέα. Είναι, είναι σαφές ότι αυτό το φαινόμενο συνεισφέρει για, στην επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κόστος της μη ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας ε, ξεπερνούν τα 160 δις ε, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία. Και εδώ έχουμε και την ε, ανάγκη για την πρωτοβουλία εγγύησης για τους νέους. Είναι πολύ σημαντική η υπόθεση αυτή, ώστε η εγγύηση για τους νέους να μπορεί να διαμορφωθεί σε, ε, αποτελεσματικά πλαίσια μέσω των κονδυλίων του Κοινωνικού Ταμείου, με πολύ στενή συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, μεταξύ των εθνικών αρχών, περιφερειακών και τοπικών αρχών ε, και των υπηρεσιών προσφορά εργασίας. Το κλειδί εδώ είναι να βοηθήσουμε τους νέους μας, να τους βοηθήσουμε ώστε να μπορέσουν να βρουν τη γεφυροποίηση από τα σχολεία και την εκπαίδευση στον χώρο εργασίας, στον κόσμο της εργασίας. Πρέπει να δράσουμε και οι συστάσεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη-μέλη που ζουν και περνάνε τεράστιες δυσκολίες οικονομικές και κοινωνικές σήμερα θα πρέπει να βοηθηθούν. Διακόπτεται το μικρόφωνο από τον Πρόεδρο. Σας ευχαριστούμε πολύ αγαπητοί συνάδελφοι κυρία Μπάστος. Ακολουθεί τώρα για ένα λεπτό η συνάδελφος κυρία Στάινρουκ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, η ανεργία των νέων δεν μπορεί μόνο με κενά, κενούς λόγους και δεκάρικους λόγους να αντιμετωπιστεί. Πρέπει με κονδύλια να αντιμετωπιστεί. Το παράδειγμα της Αυστρίας δείχνει τι πρέπει να γίνει. Ως εισηγήτρια του προγράμματος για την καινοτομία, κοινωνική καινοτομία, δείχνει το τι πρέπει να γίνει ώστε αυτά τα οποία προτείνονται για την πρωτοβουλία για τους νέους στην Ευρώπη πανευρωπαϊκά να μπορέσουν να δρομολογηθούν και να είναι αποτελεσματικά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υπόψη του προγράμματα με την ανταλλαγή βέλτιστων ε, προδιαγραφών και βέλτιστων εμπειριών ε, να προχωρήσουν. Είναι ακατανόητο ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών λένε ναι, θέλουμε να καταπολεμήσουμε την ανεργία των νέων, από την άλλη όμως πλευρά δεν είναι είναι πρόθυμοι αυτή την καλή πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να την υποστηρίξουν. Και θα έλεγα ότι θα έπρεπε οι αρχηγοί κυβερνήσεων να ισχύνονται, να ντρέπονται, διότι καινούς δεκάρικους λόγους εκφωνούν χωρίς να ακολουθούν πράξεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρος, σας ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Στάινρου. Για ένα λεπτό, ο κύριος Γκουτιέρες Πριέτο, παρακαλώ. Κύριε Άντορ όσο θα διαρκέσει η παρέμβασή μου θα έχουν χαθεί δύο θέσει εργασία στην Ισπανία. ένα νέο μάλιστα θα είναι αυτό που θα χάσει την εργασία του. Και αυτό συμβαίνει σε πολλέ χώρε τη Ένωση. Και εσεί, όσο συμβαίνουν αυτά, δεν έχετε καταφέρει να δρομολογήσετε ούτε μία πρόταση, ένα πρόγραμμα για να αλεξιτοποιήσετε αυτό το πρόβλημα, την κατάσταση που αντιμετωπίζουν χιλιάδε πολίτε. Άρα, πρώτον, έρχεται αργά αυτό το μέτρο. Όσο γίνονται όλα αυτά όμως εσείς δεν μπορείτε να δρομολογήσετε ένα φιλόδοξο συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, κάτι που ζητά το Κοινοβούλιο και αναφέρεται ζητήματα κουρικότητα, αρμοδιοτήτων, δημιουργώντα μεγαλύτερη απελπισία και μεγαλύτερη απογοήτευση. Γιατί η Ευρώπη σήμερα, κύριε Επίτροπε, εξακολουθεί να έχει ε, πόρου. 10% ε, των κονδυλίων που έχουν εγγραφεί στον προπολογισμό αλλά δεν ε, χρησιμοποιήθηκαν στην Ισπανία φέτο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αυτή την εγγύηση για την νεολαία. Οι τράπεζε που έχουν πόρου όμω ε, ε, είναι πάρα πολύ σφιχτέ και δεν δίνουν χρήματα στου νέου. Λοιπόν, κόβεται το μικρόφωνο. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε πολύ συνάδελφε Γκουτιέρε Πρίετο. Ακολουθεί για ένα λεπτό ο συνάδελφο κύριο Χάουιτ, παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι το 40% των Βρετανών κάτω των 25 ετών είναι άνεργοι. Μολονότι υπάρχει ένα πρόγραμμα βρετανικό το οποίο υποτίθεται ότι θέλει να βοηθήσει τους νέους, ωστόσο ελάχιστος καλύπτει. Και ξέρετε ότι ε, πολύ συχνά μέσω της φορολογίας προσπαθούν να βρεθούν οι απαραίτητοι πόροι για να χρηματοδοτούν τέτοια προγράμματα υπέρ των νέων. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι στην περιοχή της Ανατολικής Αγγλίας, στην οποία εκπροσωπώ, είναι η δεύτερη περιφέρεια η οποία πλήττεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ανεργία των νέων. Και από ό,τι φαίνεται η κατάσταση αυτή θα επιδεινωθεί. Ένα στου πέντε νέου στην περιοχή μου λέει ότι έχουν καταστραφεί εντελώ οι προοπτικέ του. Άλλοι θεωρούν ότι πλήττονται εντελώ από κατάθλιψη. Η Έμιλι, μια κοπέλα από τον Νόρφορκ, χρειάστηκε στην ηλικία των 13 ετών να φύγει από το σχολείο. Είχε πεθάνει ο πατέρα τη και αυτή τη στιγμή υποφέρει από κατάθλιψη. Αντί για χάπια, σα δώσουμε ελπίδα. Σα ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφε Χαόι. Για ένα λεπτό, η συνάδελφο κυρία Νεβεντάλοβα. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, χαίρομαι που και πάλι ξανασυζητάμε την κατάσταση στην Ευρώπη. Την ξανασυζητάμε, διότι η κατάσταση εξακολουθεί να παρουσιάζει ένα μείζον πρόβλημα για μας. Καλωσορίζω την πρόταση του Επιτρόπου Άντο για την εγγύηση για την νεολαία. Καλωσορίζω το γεγονό ότι ήταν μια σοσιαλιστική πρωτοβουλία αυτή. Μια πρωτοβουλία του κόμματο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών ώστε εμπνεύστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από ιδέες της αριστεράς. Είναι πολύ σημαντικό για τους νέους να τύχουν κατάρτισης, μιας μαθητείας, μιας δυνατότητας άσκησης ως μαθητευόμενων. Είναι μια δυνατότητα να βρουν μια διέξοδο από αυτό το πρόβλημα. Οι νέοι είναι το μέλλον μας στην Ευρώπη. Πρέπει να επενδύσουμε στο μέλλον μας επενδύοντας στους νέους. Τα κράτη-μέλη δεν έχουν πια χρήματα και όμως 10 δις ευρώ επαρκούν για να δημιουργηθούν 2 εκατομμύρια θέσεων απασχόλησης για τους νέους. Χρειαζόμαστε κάτι περίπου σαν 30 δις ευρώ για να μπορέσουμε να απασχολήσουμε όλους τους σήμερα άνεργους νέους. Αν επενδύσουμε σε αυτούς τους νέους ανθρώπους θα έχουμε κάτι παραπάνω από κερδοφόρα επιστροφή από αυτή την επένδυση που θα κάνουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφε Νεβεντάλοβα. Για ένα λεπτό Στη συνέχεια Γκάρδια Σαμπάρ Ρουμπιάλ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, καταπολέμηση της ανεργίας των νέων είναι τμήμα των γραμμών δράσης της Κομισιόν, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, όπως τις εγκρίναμε στο πλαίσιο για την Ευρώπη το 2020. Έχουμε τη μεγαλύτερη νεανική ανεργία από το 1995. Επομένως, οποιαδήποτε πρωτοβουλία θα είναι καλοδεχούμενη. Ωστόσο, αυτή η πρωτοβουλία ότι δηλαδή οποιοδήποτε νέος θα μπορεί να έχει τη δυνατότητα να βρει μια θέση ε, εργασίας ε, είτε για να σπουδάσει κάτι ακόμη ή για μια άσκηση μετά από τέσσερι μήνες ανεργίας. Έχει κάποιου περιορισμού. πρώτα γιατί τι γίνεται με τους ε, κάτω των, των, των 25 και τι γίνεται με τη χρηματοδότηση που δεν είναι συγκεκριμένη. Γι' αυτό ζητάμε να ανεβάσετε την ηλικία στους, στα 30 έτη να έχετε σαφή κριτήρια για όλα τα κράτη-μέλη, ώστε να υπάρχουν ποιοτικέ απαιτήσει, παραδείγματο χάρη, ε, σε ό,τι αφορά τι προποθέσει ε, για την πρόσληψη. Και στα επόμενα 7 χρόνια θα πρέπει να διαθέσετε επίση επαρκή χρηματοδότηση για αυτή την πρωτοβουλία. Σα ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφε Γκάρδια Σάβαρ Ρουμπιάλ. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στη διαδικασία είναι εξαιρετικά δύσκολο τώρα αυτό. Έχουμε 20 που ζήτησαν τον λόγο να παρέμβουν για ουσιαστικά 5 όλα και όλα λεπτά. Και πέρα από αυτό έχουμε και το πρόβλημα ότι πολύ λίγοι συνάδελφοι ήταν πειθαρχημένοι. Έπρεπε να αφαιρέσω τον λόγο, να κόψω το μικρόφωνο από τρει συνάδελφους. Γι' αυτό αποφάσισα να κάνω το εξή. Να προτείνω συνάδελφοι, δεν θα ληφθεί κανεί υπόψη που σε αυτή τη συζήτηση προηγούμενα παρενέβη. Και στην προηγούμενη συζήτηση υπό αυτό το θέμα μπόρεσε να παρέμβει διότι στην προηγούμενη συζήτηση όποιος έλαβε τον λόγο δεν θα παρέμβει στη συζήτηση Καστιάη. Ελπίζω να συμφωνήσετε όλοι, δεν μπορώ να το αλλάξω αυτό. Δεν θα υπαρκέσει ο χρόνος. Πρώτος θα λάβει τον λόγο η συνάδελφος κυρία Μάτσε Κούκοβιτς, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι η εγγύηση για τους νέους, για την νεολαία είναι κάτι το οποίο καλοχαιρετίζω, είναι ευπρόσδεκτο και αυτό γιατί, διότι οι νέοι οι οποίοι δεν έχουν εργασία δεν μπορούν να ιδρύσουν οικογένεια, να κάνουν οικογένεια, δεν μπορούν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και ούτε μπορούν τη δημιουργικότητά τους να την εκμεταλλευτούν και την, να την αναπτύξουν. Και γι' αυτό επιπρόσθετη κατάρτιση απαιτείται, παράδειγμα για την ψηφιοποίηση, ε, για τον κόσμο τον ψηφιακό δυνατότητα να βρουν απασχόληση μετά από τέσσερις μήνες για παράδειγμα ανεργίας, περίοδου ανεργίας. Αυτό θα ήταν ευκταίο και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το ευρωπαϊκό αυτό πρότυπο να μπορέσει να επικεντρωθεί στους νέους, στην νεολαία. Όμως εδώ βλέπουμε ότι η λύπη απουσιάζει, απουσιάζουν τα κίνητρα και τα ερεθίσματα. Δεν είναι σαφές ότι όλα αυτά θα στεφτούν με επιτυχία στο τέλος τέλος αν δεν τονίσουμε το ότι οι νέοι είναι ένα μέρος της λύσης και όχι ένα μέρος του προβλήματος μόνο. Ευχαριστούμε πολύ συνάδελφε Ματσέη Κούκοβιτς. Στη συνέχεια συνάδελφος κυρία Σένα Λόβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί να χάσει μια ολόκληρη γενεά νέων τα ποσοστά ανεργίας των νέων πραγματικά είναι, μας ε, τρομοκρατούν τα επίπεδα ανεργίας ε, των ε, νέων ανέρχονται σε 55 και παραπάνω της 100 σε κάποιες χώρες. Έχουμε εκατομμύρια άνεργους νέων. Ε, είναι στον αθό της ηλικίας τους αυτοί οι νέοι που θα έπρεπε και θα μπορούσαν να είναι παραγωγικοί. Δεν μπορούμε να σταυρώσουμε τα χέρια και να περιμένουμε να υπάρξει οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη. Θα είναι υπερβολικά αργά αν κάνουμε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό οι πολιτικές λιτότητας και περικοπών, περικοπών ιστοδιειναικές καθ καθιστούν τα πράγματα ακόμα πιο επώδυνα και δυσχερή. Και καλωσορίζω ιδιαίτερα την πρόταση για ένα πρόγραμμα εγγύησης, εγκυοδότησης των νέων. Είναι επίγουσα η κατάσταση, πρέπει να δράσουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό το μέσο να ενταχθεί σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και να συνειφανθεί με τις δικές τους προσπάθειες, ώστε όλοι να ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Στη συνέχεια, Κρόμπεργκ, παρακαλώ. Η Φιλανδία έχει μια πολύ καλή εμπειρία με την εγγύηση για τους νέους. Ένα 80% των ανέργων έχουν χρησιμοποιήσει την εγγύηση αυτή. Οι περισσότεροι νέοι έχουν καταφέρει να πάρουν καλύτερες αποφάσεις μετά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό και έχουν βελτιωθεί επίσης και οι υπηρεσίες σχετικές με την ανεργία. Προκειμένου όμω να καταφέρουμε να υποστηρίξουμε αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, θα πρέπει να έχουμε και πραγματικές θέσεις εργασίας. Αν δούμε το νότο της Ευρώπης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει και μία μετακίνηση των εργαζομένων ανάμεσα στις διαφορετικές χώρες στα πλαίσια της εγγύησης για τους νέους, έτσι ώστε νέοι από την Ισπανία να μπορούν να εργαστούν για παράδειγμα στη Γερμανία. Αν τελικά χρηματοδοτηθεί από τα διορθωτικά ταμεία η πρωτοβουλία αυτή, είναι πολύ σημαντικό τα ταμεία αυτά να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν, προκειμένου να βρουν δουλειά και κάποια άτομα στι υπηρεσίε απασχόληση. Διαφορετικά δεν θα έχει καμία απολύτω αξία αυτή η εγγύηση για του νέου. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μάρφη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ καλά εκφράζει την λύπη της η Κομισιόν ε, για την κρίση και την ενεργεία των νέων. Αλλά γιατί έχουμε αυτή την κρίση, δεν διαρωτηθήκατε. Αυτό ε, δεν οφείλεται στο ότι δεν είναι αρκετά σπουδασμένοι, δεν έχουν εργασιακή εμπειρία ή δεν είναι ευέλικτοι νέοι, αλλά οφείλεται στην πολιτική λιτότητα της Κομισιόν, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της πλειοψηφίας των μεγαλύτερων πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου αν δεν υπάρξουν μαζικέ δημόσιε επενδύσει, αυτή η εγγύηση για την ΕΛΕΑ θα είναι μια κενή υπόσχεση ακόμη. Είναι ένα πρόσχημα ε, τότε για να έχουμε μέτρα όπως ε, ε, κάποια μέτρα τα οποία θα δημιουργήσουν μια σειρά φτηνού εργατικού δυναμικού ενώ οι νέοι σε όλη την Ευρώπη πρέπει να κινητοποιηθούν και να ζητήσουν δράση τώρα για να βρουν θέση θα πρέπει λοιπόν να έχουμε επενδύσει δημόσιες και τεπτοβάθμια εκπαίδευση με ελεύθερη πρόσβαση σε όλους. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σαραβράκος για το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε και συνάδελφοι, καταχνιά, λιτότητα, ανεργία και κατάθλιψη πάνω από την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο οικονομικό θέμα η ενεργία είναι προεχόντως ψυχιατρικό. Οδηγούμε σε ψυχική ανομαλία μία ολόκληρη νέα γενιά. Κατόπιν τούτου χαιρετίζω και δεν μπορώ αλλιώς να κάνω με τη σειρά μου την πρωτοβουλία για τη συζήτηση αυτής της υποθέσεως. Τα σχέδια για τα προγράμματα εγγύησης για τους νέους πρέπει να προχωρήσουν κύριε Επίτροπε. Δεν πρέπει να μείνουν μια πρωτοβουλία στα χαρτιά και στις λέξεις. Είναι απαραίτητο να καταλάβουμε ότι τα μέτρα λιτότητος πάνω από την Ευρώπη και η ανεργία των νέων, των μορφωμένων νέων, δημιουργούν ένα νέο επιστημονικό προλεταριάτο που θα μας πνίξει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Στόγενοφ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Παρεμβαίνω ω ο νεότερο σε αυτό το κοινοβούλιο και προέρχομαι και από ένα κόμμα που τα μέλη του 80% είναι νεότερα από 30 ετών. Δεν θα ήθελα να υπάρξουν περισσότερες γενικές ε, δηλώσεις ή τοποθετήσεις, γι' αυτό θα αναφερθώ σε ένα πολύ συγκεκριμένο εξειδικευμένο πρόβλημα. Πολλές από τις επιχειρήσεις απαιτούν και ζητούν οι νέοι να, που ξεκινούν να εργάζονται να έχουν προηγούμενη πείρα. Ερώτησή μου, πώς μπορεί κάποιος που μόλις έχει βγει από ένα πανεπιστήμιο ή μια σχολή μπορεί να έχει ήδη προηγούμενη πείρα. Ένας νέος έτσι λοιπόν δεν μπορεί να βρει απασχόληση επειδή δεν έχουν λέει εντός εισαγωγικών πείρα. Δεν έχουν πείρα όμως επειδή δεν μπορούν να βρουν απασχόληση απασχόληση. Φαύλος κύκλος. Γι' αυτό απευθύνω ε, ε, έκκληση προς εμάς, Επίτροπε, να υπάρξουν τα κονδύλια εκείνα ώστε να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης για τους νέους. Και σε αυτό το εγχείρημα δεν θα έπρεπε να απαιτείται να έχουν προηγούμενη επαγγελματική πείρα, εργασιακή πείρα, διότι αυτό είναι αρνητική διακριτική μεταχείριση ει βάρο του. Και ποτέ δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε του στόχου για του οποίου κάνουμε λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Λουκατσεύσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι ε, όπως οι χορτασμένοι δεν μπορούν να καταλάβουν αυτούς οι οποίοι πεινάνε, κατά τον ίδιο τρόπο οι άνθρωποι που έχουν δουλειά δεν μπορούν να καταλάβουν τους άνεργους. Έχει έρθει κατάλληλη στιγμή προκειμένου να αρχίσουμε να εξετάζουμε πραγματικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνεργοι. Πάρα πολλέ συζητήσει έλαβαν χώρα, είδαμε πάρα πολλέ πρωτοβουλίε. Ωστόσο, οι νέοι άνεργοι εξακολουθούν και περιμένουν. Περιμένουν μία θέση εργασία. Περνάνε τα χρόνια και αυξάνουν το αριθμό τους. Η πρωτοβουλία για την εγγύηση των νέων είναι σαφώς καλή, τη χαιρετίζουμε, αλλά παραμένει απλώς πρωτοβουλία αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να λειτουργήσει στην πράξη. Μπορεί ο Επίτροπος να μας εξηγήσει πώς τα κράτη-μέλη θα αυτή την πρωτοβουλία. Δεδομένου ότι η πρωτοβουλία αυτή παίρνει απλώς τη μορφή μιας σύστασης. Αν τα κράτη-μέλη δεν αρχίσουν να εφαρμόζουν αυτή την εγγύηση για τον νέων, θα προβλεφθούν κάποιες κυρώσεις, ή ουσιαστικά δεν θα προβλεφθεί τίποτα στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ, Σιβριέσκα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η σύσταση του Συμβουλίου για την εγγύηση για την νεολαία για τους νέους μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα δώσει μια δυνατότητα στα κράτη-μέλη σε αυτό το πεδίο. Υπάρχουν όμως αρκετά ερωτηματικά σε σχέση με το τι μπορεί να γίνει σε σχέση με τη φάση εφαρμογής. Σε κάποιες χώρες απαιτείται πολύ περισσότερος χρόνος από ότι για παράδειγμα τέσσερις μήνες για κάποιον νέο να βρει δουλειά να βρει θέση απασχόληση. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ουσιαστικά ότι δεν υπάρχουν δουλειέ για αυτούς τους νέους. Περικοπές λοιπόν των δημοσίων κονδυλίων θέτουν επιπλέον προβλήματα. Δυσχεραίνουν την κατάσταση Χωρί ε, του εμπλεκόμενους ε, στην αγορά εργασία που πρέπει υποχρεωτικά να συνεργαστούν με του ανέργου για να διασφαλιστεί φυσικά η κατάρτισή του και η προοπτική εξέβρεση θέση απασχόληση για αυτού. Πρέπει να δράσουμε συντονισμένα για αυτούς που χρειάζονται βοήθεια, κανείς δεν πρέπει να υποστεί αρνητικές συνέπειες, για παράδειγμα νέες μητέρες που θα πρέπει να επιστέψουν στην αγορά εργασίας μετά τον τοκετό. Ευχαριστώ. Για κονσάρι. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, στην ιστορία, την ευρωπαϊκή ιστορία, νομίζω για πρώτη φορά αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου καλά καταρτισμένοι και εκπαιδευμένοι νέοι υποχρεούνται μαζικά να υποστούν την ανεργία, ένα καθεστώς ανεργίας. Αυτό είναι πραγματική τραγωδία. Υπάρχουν κάποιες ε, προοπτικές, ε, όμως φοβούμε ότι οι νέοι από στην μία εξάσκηση η μαθητεία θα περνάνε στην άλλη ώστε να καταρτίζονται διαρκώς όλο και καλύτερα με περισσότερα προσόντα χωρίς να βρίσκουν δουλειά. Το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε όταν περικόπτουν τα κράτη-μέλη τα κονδύλια. Για παράδειγμα και στην έρευνα και στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Και όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και εκείνη προβαίνει σε περικοπές κονδυλίων. Ε τότε τι μπορούν να κάνουν επιπλέον οι νέοι όταν η κατάρτιση μέσω αυτών των κονδυλίων που περικόπτουν ουσιαστικά ευνουχίζεται. Αν θέλουμε πραγματικά να δημιουργηθούν νέε θέσει απασχόληση, πρέπει να μεριμνήσουμε ποιοτικά υψηλό, υψηλού επίπεδου θέσει εργασία να δημιουργηθούν. Ευχαριστούμε, Ιρικόιν. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα. Όλοι γνωρίζουμε και το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές ότι χωρίς νέους δεν υπάρχει μέλλον. Αυτό το οποίο είναι αφόρητο και το είπαν και πολλοί συνάδελφοι είναι να βλέπουμε ότι έχουμε μια καλύτερα, την καλύτερα εκπαιδευμένη, προετοιμασμένη γενιά που δεν μπορεί να αναπτύξει όμως τα ταλέντα της και ότι η Ευρώπη δεν είναι σε θέση να δώσει μια συνεκτική αποφασιστική απάντηση. Συγχαίρω τον κύριο Άντορ για την πρότασή του. Όμως, πρέπει να υπάρξει και απαιτούμενη επαρκή χρηματοδότηση για να έχουμε αποτελέσματα και για να τεθεί ένα τέρμα σε αυτή την κατάσταση. Οι πολίτε δεν αντέχουν άλλε προτάσει που δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει να έχει λοιπόν του απαραίτητου οικονομικού πόρου για να είναι χρήσιμο και αποτελεσματικό για την εφαρμογή αυτή τη εγγύηση για την νεολαία. Αλλά πρέπει να πάμε και πιο μακριά. Κύριε Επίτροπε, είναι επίγουσα η κατάσταση με την ανεργία και αυτό μα υποχρεώνει να δράσουμε τάχιστα χωρί καθυστέρηση. Και όπω πάντα έρχονται πολύ αργά οι αποφάσει. Α μην γίνει το ίδιο και τώρα. Θα έχετε τη στήριξη του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ do you accept blue card? Δέχεστε γαλάζια κάρτα, μπλε κάρτα δέχεστε. Κυρία Ριγκόγεν, δέχεστε, ωραία. Παρακαλώ, η συνάδελφος Τσικάου. Σας ευχαριστώ θερμά. Επιτρέψτε μου να θέσω το εξής ερώτημα στην αξιότιμο συνάδελφο. Η ανεργία των νέων είναι μόνο τα στοιχεία αυτά, τα αριθμητικά στοιχεία αρνητικά. Πρέπει και εκείνοι που διακόπτουν τη σχολική τους εκπαίδευση και εγκαταλείπουν τα σχολεία και αυτό να μας ανησυχεί. Διότι και αυτό το ποσοστό νέων και η ανεργία των νέων <clears throat> δημιουργούν κινδύνους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τα κράτη-μέλη. Πρέπει να διασφαλίσετε όχι μόνο ότι θα είναι υψηλού επίπεδου η εκπαίδευση και κατάρτιση για τους νέους, αλλά και οι νέοι να έχουν θέσεις απασχόλησης. Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης σημαντικότατη υπόθεση Ευχαριστώ. Βεβαίω, φυσικά και συμφωνώ με τη συναδελφό μου. Αληθεύει ότι πολλοί είναι οι νέοι που εγκατέλειψαν τις σπουδέ τους λόγω των, ε, της κατάστασης στην αγορά εργασίας επειδή μπορούσαν γρήγορα να βρουν μια δουλειά που θα του έδινε χρήματα. Τώρα αυτοί οι νέοι όμω ε, πολλές φορές ε, γυρίζουν πίσω ε, στα θρανία και είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να πάρουν τα παρέτα προσόντα, να τελειώσουν τι σπουδέ τους. Αλλά πιο σημαντικό είναι να δημιουργήσουμε θέσεις εργασία όταν επανέλθουν οι νέοι αυτοί δηλαδή, στην να βρουν μια δουλειά. Ευχαριστούμε κύριο Σκέλλερ. Σας ευχαριστώ. Σε κάποιες περιοχές, περιφέρειες της Ευρώπης κάθε ένας ή κάθε δεύτερος κάτω από 25 δεν έχει ούτε θέση κατάρτισης ούτε θέση απασχόλησης. Αλλά υπάρχουν και άλλες περιφέρειες στην Ευρώπη όπου είναι οι νέοι που λείπουν από αυτές. Σε τέτοιες περιφέρειες ε, τουλάχιστον κάποιοι νέοι από κάπου αλλού θα μπορούσαν να έχουν κάποιες προοπτικές. Αλλά γι' αυτό δεν χρειάζονται δεκάρικοι λόγοι, αλλά ενημέρωση, πληροφόρηση, προσέλκυσή τους, γλωσσικά μαθήματα γλώσσας, κατάρτιση και τα συναφή. Πρακτικά μέτρα δηλαδή που πρέπει να υλοποιούνται στα κράτη-μέλη προ αυτήν την κατεύθυνση και που σε ένα χειροπιαστό παράδειγμα μπορούν να είναι έκφραση ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Διότι αν χαθεί μια ολόκληρη γενεά, αυτό δεν είναι μόνο πρόβλημα και κακό, αρνητικό στοιχείο για την οικονομία, είναι τεράστιο πρόβλημα για την κοινωνία και τη δημοκρατία μα συνολικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Πάσκα. Ευχαριστώ, πρόεδρε, κύριε, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Δεν ότι λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να δημιουργήσει θέσεις εργασία για του νέου, αλλά θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σα την εμπειρία που έχω από τη δική μου τη χώρα. Μολονότι οι συνθήκε είναι πάρα πολύ δύσκολε, η χώρα μου γνωρίζει αυτή τη στιγμή μια οικονομική ανάπτυξη. Υπάρχουν ε, ορισμένες εταιρείες ηλεκτρονικών προϊόντων, καθώς επίσης και η αυτοκινητομηχανία χρειάζεται νέους εργαζόμενους. Ένα 25% των νέων είναι άνεργοι. Ωστόσο όμως οι νέοι μας δεν ενδιαφέρονται για αυτές τις θέσεις εργασίας και αυτό γιατί δεν έχουν την κατάλληλη κατάρτιση για αυτές τις θέσεις εργασίας. Οι περισσότεροι σπουδάζουν ανθρωπιστικές επιστήμες οι οποίες δεν αξιοποιούνται ιδιαίτερα καλά στη βιομηχανία στη συνέχεια. Μέρο λοιπόν του προβλήματο ενδεχομένω να είναι η αναντιστοιχία ανάμεσα στα πανεπιστημιακά πτυχία και προγράμματα και την εργασία που μπορεί να προσφέρει μια επιχείρηση τη σημερινή ημέρα. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κράτσα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, σε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που ακούστηκαν από τους συναδέλφους θα ήθελα να συμπληρώσω ότι η κατάσταση είναι επίγουσα γι' αυτό απαιτούνται μέτρα ε, άμεσα και αποτελεσματικά για να αποφύγουμε την αύξηση της ανεργίας η οποία έχει αυτή την τάση σε όλες τις χώρες όχι μόνο στις χώρες του νότου όπως είναι η χώρα μου αλλά και ε, σε πολλές χώρες του κέντρου ε, ε, που ανθίστανται καλύτερα σήμερα και τη φυγή των νέων από την ευρώπη όχι μόνο από τη χώρα τους από την ευρώπη με ό,τι σημαίνει αυτό για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Ε, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να ληφθούν άμεσα λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη έχουμε προγράμματα για την νεολαία ήδη έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αξιολόγηση ουσιαστική και σοβαρή ούτως ώστε να πάρουμε τα καλύτερα συμπεράσματα για να αξιοποιήσουμε και να αποφύγουμε τα λάθη και την κατασπάταληση πόρων που δεν απέδωσαν τα δέοντα. και από την άλλη πλευρά ήθελα να τονίσω ότι αν δεν υπάρξει ένα ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης στις χώρες του νότου Η ισορροπία μεταξύ των χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης δεν θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για βιώσιμη ανάπτυξη και σταθερότητα που αυτές θα φέρουν επενδύσεις απασχόληση και συγκράτηση των νέων στις χώρες τους και στην ευρώπη. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Κέλλη. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και πάνω από όλου, ε, λόγω της οικονομικής ύφεσης έχουν πληγεί νέοι που πηγαίνουν στο σχολείο, σπουδάζουν, ε, μελετούν σκληρά, ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, προετοιμάζονται, κάνουν μεταπτυχιακά και μετά δεν βρίσκουν δουλειά. Υπάρχουν σπουδαστές οι οποίοι πάνε τρεις-τέσσερις ώρες ε, συνεντεύξεις και μετά ε, δεν, κάνε, δεν ακούν καν τίποτα. Δεν παίρνουν κανένα, καμιά απάντηση. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε σοβαρά το πρόβλημα και οι νέοι που δεν βρίσκουν θέση εργασία δεν θα πρέπει τελικά να πάθουν κατάθλιψη. Επίσης έχουμε το φαινόμενο της μετανάστευση, όπως στη χώρα μου όπου ε, υπάρχουν ε, χάρη μέχρι από, από να έχουν μείνει τρεις μόνο στη χώρα και όλοι οι άλλοι να έχουν φύγει. Λοιπόν, θα πρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα επιγόντως. Ε, Ευχαριστούμε. Ολοκληρώθηκε η δικασία Catch the Eye. Επομένω, το λόγο τώρα έχει ο Επίτροπος Άντορ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, ήταν πολύ σημαντική συζήτηση για ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να αποτελέσει μια εμβληματική πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σε αυτή την ε, τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο. Η Ιρλανδική Προεδρία ξεκίνησε και την προηγούμενη εβδομάδα στο Δουβλίνο. Ε, είδαμε ότι δεν είναι για τον Υπουργό μόνο πρωτοβουλία αυτή μια προτεραιότητα, αλλά και για όλη την Ιρλανδική κυβέρνηση. Αυτό έχει σημαντική, έχει μεγάλη σπουδαιότητα γιατί το Συμβούλιο των Υπουργών Απασχόλησης θα πρέπει πράγματι το Φεβρουάριο να ε, συμφωνήσει για να μπορέσουν ε, να ξεκινήσουν ε, τα μέτρα για την εφαρμογή το στο δυνατό αυτής της πρωτοβουλίας. Ξέρουμε ότι είναι πολύ σοβαρή κατάσταση. Επειδή όμως άκουσα κάποια ζητήματα που αφορούσαν την Ιρλανδία και την Ισπανία, κάποιοι συνάδελφοι σας δηλαδή καταλογίζουν ε, την ευρωπαϊκή πολιτική που ασκείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να σας πω ότι πρέπει να το μελετήσουμε πιο σοβαρά το θέμα. Εγώ είμαι ανοιχτό πάντοτε στη συζήτηση και μπορούμε να συζητήσουμε τα αίτια της απαρχίας αυτής της κρίσης. Ε, αλλά είναι λίγο σκληρό να πει κανείς ότι φταίει η ευρωπαϊκή πολιτική. Είχαμε στην Ιρλανδία ένα ε, σύστημα τραπεζικό ε, που είχε χτιστεί στην άμμο. Αυτό, γι' αυτό δεν φταίει η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Πολιτική. Ούτε η φούσκα των ακινήτων που έσκασε στην Ισπανία είναι στέξιμο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή κάποιου άλλου θεσμικού οργάνου. Ξέρω πώ έχει κατάσταση σήμερα, είναι πάρα πολύ σοβαρή και μάλιστα προχθέ κάναμε Σεπτεμβρίου μία ε, πρόταση και συζητούσα από χθε λοιπόν με ένα συμβούλιο νεολαία στην Ισπανία και θα ξαναεπισκεφθώ εντό του Ιανουαρίου την Ισπανία και πρέπει να πω ότι σίγουρα επλήγει περισσότερα από όλε τι άλλε από την ανεργία των νέων, αλλά γενικώ ε, τα ποσοστά τη ανεργία είναι τα χειρότερα στην Ισπανία. Αυτή λοιπόν η πρωτοβουλία για την εγγύηση για την νεολαία δείχνει ε, το καλύτερο πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ανταλλαγή καλύτερων πρακτικών, ότι προσκαλούνται οι κοινωνικοί εταίροι να έχουν μια οικοδομική συνεργασία όλοι μεταξύ τους και επίσης ε, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ε, πλέον αποκτά ουσία. Θέλουμε λοιπόν να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως αυτές που διδαχθήκαμε τη Φιλανδία την Αυστρία. Θα μιλήσει ο Πρωθυπουργό αύριο εδώ και ελπίζω να αναφέρει υπερήφανα ε, τα θέματα αυτά και το ρόλο που διαδραμάτισε και αυτή η εγγύηση για την νεολαία στη χώρα του. Βέβαια, μόνο αυτό το μέτρο δεν επαρκεί σε εγγύησεις για την νεολαία για την καταπολέμηση της ενέργειας των νέων. Υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία, θα εφαρμοστούν και άλλε. Η διπλή κατάρτιση, παραδείγματο χάρη, έχουμε το μοντέλο τη Αυστρία ή τη Γερμανία, το είπε και ο κύριο Μαν. Τα ξέρει πολύ καλά, σίγουρα. Θα μπορούσαμε να το ε, εφαρμόσουμε και σε άλλε χώρε. Βελτίωση λειτουργία των υπηρεσιών απασχόληση επίση είναι ένα μέτρο. Πρόσβαση εργασίας, λοιπόν, πρόσβαση σε θέσεις εργασίας ε, στη χώρα αλλά και εκτός. Κινητικότητα επίσης, ένα άλλο σημαντικό τομέα που επεξεργαζόμαστε. Και βέβαια θα συνεχίσουμε σε συνεργασία με τους ευρωβουλευτές. Κυρία Χίρς, είπε πολύ σωστά ότι δεν είναι εγγύηση για θέση εργασία αυτή η εγγύηση για την όλα και δεν θα απαλείψει εντελώ την ανέργεια των νέων. Έχει όμω τη δυνατότητα να περιορίσει σημαντικά τα ποσοστά τη ανέργεια των νέων. Θα πρέπει να προσφέρει πακέτα θέση εργασία, επιμόρφωση, άλλε δηλαδή δυνατότητε επανεκπαίδευση. Και ακόμη και αν η αρχική προσφορά για κάποιον είναι μια δυνατότητα να μάθει κάτι, να καταρτιστεί, θα είναι χρήσιμη, πρέπει να είναι χρήσιμη και θα πρέπει να ε, προσθέσει στην απασχολησιμότητα του ατόμου, στο δεδομένο της χώρας ε, ή της ε, περιοχής στην οποία κατοικεί. Στο Κοινοβούλιο έχει γίνει και κατά το παρελθόν συζήτηση για το θέμα της flexicurity, ευελιξίας με ασφάλεια δηλαδή. Γιατί υπήρξε λίγο ε, να είναι χολό αυτό το μέτρο, δηλαδή πιο πολύ τονίσαμε την ευελιξία και όχι τόσο την ασφάλεια. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την απασχόληση λοιπόν για την νεολαία μας, που, τη γενιά αυτή που βιώνει δύσκολες στιγμές, αυτό είναι γεγονός. Και θα πρέπει η ασφάλεια αυτή να είναι και στο μέλλον. Δεν θα πρέπει να δώσουμε δηλαδή απάντηση μόνο ε, για την επίγουσα σημερινή κατάσταση, την κρίση, αλλά θα πρέπει αυτό να συνιστά και μια δομική βελτίωση για τη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Ιδίω για τη μετάβαση από το σχολείο στην δουλειά, στη θέση εργασία. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, όπω είπα και στην εισαγωγική μου ομιλία, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Οι πόροι όμω πρέπει να ιεραρχηθούν κατά προτεραιότητα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Και τώρα, αλλά και για ε, το μέλλον, το απότερο. Φυσικά και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που άκουσα στη συζήτηση. Αρκετά κροκοδίλια δάκρυα έχουν χυθεί για την ανεργία στην Ευρώπη. Τώρα αυτό που χρειάζεται πλέον είναι σαφής ε, παρέμβαση. χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του τρέχοντος έκτα, αλλά και για το επόμενο ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό θα είναι το κλειδί για να στηριχθεί οικονομικά η εγγύηση για την νεολαία. Σε ό,τι αφορά τώρα συγκεκριμένα project, η κυρία Κοστέλο ρώτησε, τα σχετικά για την Ιρλανδία θα τα διευκρινίσουμε τι επόμενε εβδομάδε. Το Φεβρουάριο, ε, αν χρειαστεί, θα μεταβώ δύο φορέ στην Ιρλανδία για να το συζητήσω το θέμα αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν όλου και όλε εσά για τη συζήτηση αλλά και για την υποστήριξή σα, όχι μόνο σήμερα αλλά και τα τελευταία τρία χρόνια. Από την αρχή από τότε που προτάθηκε η στρατηγική την Ευρώπη το 2020. Κυρία Τούρινεν, κυρία Μπερέ και πολλοί άλλοι από την Επιτροπή Απασχόληση έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Αυτή την υποστήριξη θα τη χρειαστούμε και στο μέλλον. Γιατί δεν σταματά εδώ η συζήτηση. Πρόκειται όμω για μια υποστήριξη που βλέπουμε τώρα να παίρνει αυτή η πρόταση για την εγγύηση για την ολία και θα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα είναι ένα μήνυμα προς τα κράτη-μέλη γιατί πρέπει να συμφωνήσουν και αυτά το Φεβρουάριο και για τη χρηματοδότηση βέβαια μεταγενέστερα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Έχουμε λάβει λοιπόν μια πρόταση ψηφίσματος. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη προβλέπεται κοινή συζήτηση όσον αφορά την πολιτική συνοχή σε Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκής